Welcome to the uh, Employment Committee meeting. Uh, can we work... Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε να εγκρίνουμε παρακαλώ την σε διάταξη. Ναι, από ό,τι φαίνεται, χωρίς τροποποίησεις. Μερικές ανακοινώσεις. Καταρχήν για τη διερμηνία έχουμε όλες τις γλώσσες με εξαίρεση φιλανδικά, μαλτέζικα και κροατικά. Έχουμε μάλιστα και διερμηνία ε, από και προς την νοηματική για το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική των Ατόμων με Αναπηρία. Αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης καταρχήν. Ο κύριος Ράτκε από το ΕΛΚ. Γίνεται τακτικό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης. Καλώς ήρθατε λοιπόν ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης. Και ο Σβέν Σούλτς που ήταν προηγουμένως τακτικό μέλος της Επιτροπής γίνεται αναπληρωματικό αντικαθιστώντας την κυρία Γκρέσλε. Και τέλος, ο κύριος Ρέι Φίντς από το EFTD αντικαθίσταται από την κυρία Λουίς Μπούρς από την ίδια ομάδα, EFTD, στη θέση του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Απασχόλησης. Καλώς ήρθατε όλοι. Καλή τύχη στην ανάληψη των καθηκόντων σας. Περνάμε στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και πάμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες. Έχετε μαζί σας τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Ε, we start with the amendment. Ξεκινάμε με την τροπολογία 117 τη σχεδίου έκθεση για τις πολιτικές ελάχιστου εισοδήματο ως μέσο αντιμετώπισης της φτώχειας. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Υπέρ παρακαλώ. Η κυρία Γεζοβιέσκα. Ε, λυπάμαι, αλλά έχω ξεχάσει την ηλεκτρονική μου κάρτα. Θα ψηφίσω διανατάσσω τη χειρός. Ε, δεν ξέρω τι προβλέπετε εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε. Μήπως μπορούν να σας στείλουν μία κάρτα για να ψηφίζετε. Do you get it now? από τη βλέπω σας φέρνουν μία κάρτα για την κατάσταση της δικής σας. Περνάμε λοιπόν στη ψηφοφορία της τροπολογίας 117. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Συμβαστική τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε κατευθείαν στην τροπολογία 130 ένα Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 131, μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Can we close the vote? Ψηφίσατε όλοι να κλείσουμε την ψηφοφορία. Θα χρειαστεί να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 131. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Με μία ψηφοδιαφορά. try it Άντε, τρίτη και τυχερή. Μία ακόμη επανάληψη. Θα καταμετρήσουμε και εσάς κυρία Γεζοβίετσκα στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, τρίτη και τελευταία φορά ψηφίζουμε για την 131. Ε, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε δύο συναδέλφους χωρίς κάρτες ψηφοφορίας και ζήτησαν να προσμετράτε και τις δικές τους ψήφους. Ανέκαθεν να γινόταν αυτό. Ε, δεν λέω ότι σώνει και καλά πρέπει να γίνει και τώρα, αλλά μέχρι στιγμής κάθε φορά που κάποιος ξεχνούσε την κάρτα του μπορούσε να ψηφίσει δηλώνοντας την ψήφο του. Καλώς, τρίτη φορά λοιπόν. Ψηφίζουμε για την 131 τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ποιοι δεν έχουν τις κάρτες και πρέπει να μετρήσουμε. Γκέρικε και Γιαζοβιέτσκα. Ψηφίζουν κατά και οι δύο.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 Αυτή είναι μία λύση. Η άλλη λύση είναι να αρνηθούμε τον συνάδελφο που κατέθεσε καθυστερημένο, οπότε είναι ισοπαλία. Εντάξει, αποφασίσαμε 23 ψήφοι υπέρ, 22 κατά. Κυρία Πρόεδρε. Ah, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λυπάμαι. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχει και ο εσωτερικός κανονισμός. Ε, συμπαθώ την κυρία Χάρκιν, μας είπε έτσι ήθιστε. Συγγνώμη, αλλά οι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Άλλοι θα έρθουν μετά από ένα εικοσάλεπτο και θα θέλουν να ψηφίσουν στις παρελθούσες ψηφοφορίες. Σας ζητώ να εφαρμόσετε τον κανονισμό. Πρέπει να ερχόμαστε εγκαίρως μαζί με την κάρτα ψηφοφορίας μας, η, δεμή, ο, ο, η δεν λαμβάνεται υπόψη. Παρακαλώ με βάση αυτό το, τον κανόνα και τον κανονισμό να δράσετε αναλόγως. Η κυρία Γεζοβιέσκα. Ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι εφαρμόζουμε τον εσωτερικό κανονισμό. Εναπόκειται στον Πρόεδρο να συμφωνήσει να λάβει υπόψη τις ψήφους των συνάδελφων που ξέχασαν ε, ή που δεν έχουν τις ε, κάρτες ψηφοφορίας. Νομίζω ότι δεν φταίμε εμεί που δεν έχουμε τι κάρτε. Το σημαντικό είναι η παρουσία μα, γιατί ήρθαμε για να ψηφίσουμε. Ηλεκτρονικά ή όχι δεν έχει τόση σημασία. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, μπορούμε κάλλιστα, αν το δεχτεί η πρόεδρο, να ψηφίσουμε διανατάσσεω τη χειρό. Ε, αν γίνεται αυτό που γίνεται τώρα εδώ, κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει και στην Ολομέλεια. Όποιο δεν έχει την κάρτα να σηκώνει το χέρι και να λέει είμαι υπέρ ή κατά. Δεν μπορεί να γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όποιο ξέχασε την κάρτα του, απλά δεν συμμετέχει στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. μου επισήμαναν ότι οι συντονιστές της συνεδρίασή τους συμφώνησαν όσοι δεν έχουν τις κάρτες ψηφοφορίας τους να λαμβάνονται υπόψη παρόλα αυτά στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το έχουν αποφασίσει οι συντονιστές. Ας προχωρήσουμε επιτέλου, γιατί αλλιώ θα βραδιάσουμε στην πρώτη ψηφοφορία. Ο κύριο Λαβριέ. Δύο παρατηρήσεις σύντομε. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων πολλοί συνάδελφοι είχαν ξεχάσει τις κάρτες τους και ψήφος τους ελήφθη υπόψη χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι γίνεται συνήθως. Δεν μιλάμε για ονομαστική ψήφο εδώ, δεν μιλάμε για ονομαστική κλίση. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε πώς ψηφίζουν οι συνάδελφοι. Δεν πρόκειται για ονομαστική κλίση. Όταν μιλάμε για ονομαστική κλίση, εφόσον δεν έχουμε κάρτα, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη φυσικά η ψήφος. Αλλά εδώ μιλάμε για τη γνώμη επί μίας τροπολογίας. Συνεπώς λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ε, είτε έχουμε κάρτα είτε δεν έχουμε κάρτα θα μπορούσαμε να ψηφίζουμε και με το όρθιο ή καθιστή επίσης. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Yes, we can uh, uh, have a Θα μπορούσαμε να το συζητάμε πολύ ώρα ακόμη. Χρησιμοποιώ λοιπόν τη διακριτική ευχέρεια Τη Προέδρου και θεωρώ ότι έκλεισε ψηφοφορία και το αποτέλεσμα είναι 23 ψήφοι υπέρ και 22 κατά. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες αν θέλουμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα στις επόμενες ψηφοφορίες για το ίδιο θέμα να το κάνουμε. Οπότε προχωράμε στην επόμενη τροπολογία, την 133. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 133. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, is there Μήπως έχουμε κάποιον υπεράριθμο ή κάποιον που δεν δικαιούται να ψηφίσει και παρόλα αυτά ψηφίζει. Όσοι δεν έχουν τις κάρτες τους, πώς ψηφίζουν. Μόνο για η κυρία Γιαζοβέτσκα έμεινε χωρίς κάρτα. Οκ, οπότε έχουμε ισοπαλία 22-22. Άρα απορρίπτεται η τροπολογία 133. Συμβαστική τροπολογία 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον, άντε το ελέγξουμε καλύτερα, γιατί είναι οριακή διαφορά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 18. Τέλος ψηφοφορίας. Α, ωραία, έχουμε και μεγάλη διαφορά. Κάτι που μας διευκολύνει. 24 ψηφοί, πέραν 11 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 140 θέλετε έλεγχο για την 138 πολύ ωραία έρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος για την 138 Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 138 με ξεκάθαρη διαφορά. 27 ψήφοι υπέρ. 27 ε, ψηφι κατά, συγγνώμη, 18 υπέρ. 140, ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 145. Α, όχι, έχει αποσυρθεί. Πάμε στη συμβαστική 19. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 153. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά η ψήφο σας δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 156. Έρχεται ο τεχνικός για να σας βοηθήσει. Η τεχνικός. 156. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 162. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 21 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική Συμβαστική τροπολογία 21α ως προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ λέω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 21α. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. 28 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 170. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ή μάλλον όχι. Ποιος είναι υπέρ. Επανάληψη. Κατά. Αποχές. Άντε στο ελέγξουμε καλύτερα. Τροπολογία 170 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 172 λέει η πρόεδρος. Ή μάλλον 171 διορθώνει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 172. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 173 και 174 μαζί ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική τροπολογία 22 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία 22 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Πρέπει να επαναλάβουμε την, τον ηλεκτρονικό έλεγχο για την 22. Είχαμε ένα τεχνικό σφάλμα. Συμβαστική τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πατήστε το κουμπί παρακαλώ. Το πράσινο αν είστε υπέρ, το κόκκινο αν είστε κατά, ο πρόεδρος. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ 13 κατά. Πάμε τώρα στην τροπολογία 186. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο και για αυτήν την 186. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. Τροπολογία 190. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 205. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά. Εγώ βλέπω να απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 206. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται οριακά με μία ψήφο διαφορά. 207. Κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 207. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 215. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω το αποτέλεσμα. Καλά. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για την 215. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 216. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι δεν καταλαβαίνω το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία 26. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 ψηφί. υπέρ, 18 κατά. Συμβαστική τροπολογία 27. Ποιο είναι υπέρ. Κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 225. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 233. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 234. Άρχεται η ψηφοφορία. Uh, and, ε, the vote is now closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ. 235. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε και την 235. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 29 ψήφοι υπέρ. 236. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές. Εγώ βλέπω μάλλον να έχει εγκριθεί. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο και για τη 236. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Οριακά, με μία ψηφοδιαφορά. Συμβαστική τροπολογία 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 253. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 253. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 29 ψήφοι κατά 17 υπέρ. 254. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για 255. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 256. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 266. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε 266 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας και απορρίφθηκε με μεγάλη διαφορά κιόλας η 267 η 267 υπέρ κατά Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Ελέγχουμε την 267. Έναρξη. Περά. Με δύο ψήφους εγκρίνεται. 268. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Η 269. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Η 271 με προφορική τροπολογία σοσιαλιστών. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 284 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 286 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Η 294 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίφθηκε. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Έλεγχος για την 296. Ε, Παρακαλώ, ζητείτε έλεγχος. Έναρξη. Πέρας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Η 297 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Οίκον 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Οίκον 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Οίκον 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οίκον 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται. Έλεγχος για την οίκον 7. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ. Οίκον 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οίκον 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οίκον 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για την οίκον 10. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. Οίκον 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την εικόν 11. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται με 27 ψήφου υπέρ. Εικόν 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εικόν 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εικόν 14. Μάλιστα. Έλεγχος την 14. Έναρξη. Πέρας. 31 ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. Οίκον 18. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ μου λέω ότι μάλλον απορρίπτεται. Έλεγχος, εντάξει. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Έναρξη και πέρας. Εγκρίθηκε 29 ψήφι υπέρ 18 κατά. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Εντολογικές σκέψεις. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οίκον ή ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Ελέγχουμε παρακαλώ τον 26. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 27. Και οίκον F ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 28. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται σου ζητείται για την 28. Έναρξη και πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. Η 30 καταπίπτει. Η 29 επίσης καταπίπτει. Η 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 41 υπέρ κατά Άποχες. Έλεγχος. Έναρξη για την 41. Πέρασε. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. 42 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά. Έλεγχο παρακαλώ γιατί 43. Πέρασε. Απορρίπταται 29 ψήφι κατά. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές την συμβαστική 10 παρακαλώ υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Η 75 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται θα έλεγα. Η 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Για την 77. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την ε, τροπολογία υπερθμών 77. Ψηφίζουμε και πέρας. Μία ψήφος διαφορά εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 τα Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται. Έλεγχος ζητείτε Για εικόν ΑΙ γιώτα. Έλεγχος παρακαλώ. Έναρξη. Και πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 25 ψήφοι κατά εικόν ζέι Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Οίκον κάπα, και υπέρ. Ε, την και κ παρακαλώ, κάπα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οίκον μη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οικονομικρον, έλεγχος για την οίκον M, μη. Μάλιστα, ηλεκτρονικός έλεγχος. Και πέρας τώρα. απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Οίκον ομικρόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την οίκον ομικρόν. Ενδεχομένω να έχουμε και το ίδιο αποτέλεσμα και πέρα στι ψηφοφορία 21 μία ψήφη υπέρ, λέει ο πρόεδρο. Οίκον πι, ρο, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος ζητείται. Έναρξη ψηφορίας και πέρας. Εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ οίκων πί, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα. συγγνώμη. Εικον Q, στην Q είμαστε. Την εικον Q, υπέρ. Κάτα. Αποχές. Ε, απορρίφθηκε. Για την εικον Q παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος έναρξη. Και πέρας. Εγκρίθηκε με 29 ψήφους Εικον U, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οίκον Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την οίκον Β. Όλοι υπέρ. Πέρας. τέσσερις υπέρ η ψήφη. Ωραία. Να περάσουμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 και 8 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Έπρεπε να τι έχουμε ψηφίσει μαζί, εν πάση περιπτώσει ψηφίσουμε ξεχωριστά. 12 υπέρ. Για την 12 παρακαλώ υπέρ. να κοιτάξουμε την 13. 13 λοιπόν, υπέρ. Τη 13 και με 14 μαζί. 13 και 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την 13 και 14 από κοινού. Έναρξη και πέρας πληροφορίας. εγκρίνονται με 10 ψήφους διαφορά. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τα έλεγα. Εντάξει, ας ελέγξουμε για την 16. Έναρξη για την 16. Πέρασε. 28 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται θα έλεγα. Ας ελέγξουμε τα 18 αν θέλετε. Έναρξε. Και πέρασε. εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. Να περάσουμε τώρα στο 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οίκον G υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε στο σχέδιο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Με νέα ονομαστική κλίση παρακαλώ. Για το σχέδιο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Πέρασε. Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ, 7 κατά και τέσσερις αποχές. Ευχαριστούμε την εισηγητρία. Και έτσι λοιπόν περνάμε στην επόμενη έκθεση. Uh, Η έκθεση της κυρίας Τόμ για τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης. Θα ξεκινήσουμε με την συμβιβαστική υπαριθμόν 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Είπαμε συμβιβαστική υπαριθμόν 3. Yeah. Those in favor. Ξανά υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 41. Α, για μια στιγμή. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 57 υπέρ κατά αποχές απερίφη να υπάρξει έλεγχος λοιπόν για την 57 ψηφίζεται πέρας απερίφη 58 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 68 πρώτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Ποιοι είναι υπέρ της ονομαστικής κλίσης τότε, σηκωθείτε παρακαλώ. Για την 68. Εντάξει, έχουμε 11. Ήσασταν περισσότεροι από 11, οπότε έχουμε ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 68, το πρώτο τμήμα. Ψηφίζεται. Επαναλαμβάνω, 68 πρώτο τμήμα, πέρα στις ψηφοφορίες, 40 υπέρ. Τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Όχι, έχει καταπέσει πλέον το δεύτερο τμήμα, λέει η Πρόεδρος. Είναι περίπου η ίδια διατύπωση. ή μάλλον υπάρχει έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Υπάρχει αντίρρηση. Μα είπα ότι έχει καταπέσει λέει η πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε λοιπόν και για το δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση πάντα στην τροπολογία 68. Ψηφίζετε παρακαλώ. Απεριφθεί 24 κατά 17 υπέρ. Τρίτο τμήμα. Καταπίπτει λέει πρόεδρος αλλά συνεχίζει λέγοντας όχι δεν καταπίπτει τελικά. Το ίδιο θα ψηφίσουμε λοιπόν για το 3 με ονομαστική κλίση μετά από αίτημα των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Ψηφίζεται. Ονομαστική κλίση για το τρίτο τμήμα της 68. Τέλος. Απερίφθη. 69. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 73. Τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος τότε για το δεύτερο τμήμα της τοπολογίας 73. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 24 κατά 18 υπέρ. Περνάμε τώρα στην 75. Προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Θέλετε να ακούσετε την προφορική τροπολογία. That means that we vote on the uh, original uh, uh, amendment. On amendment 75, those in favor. Λοιπόν, 75. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη θα έλεγα η 75. Α, έλεγχος λοιπόν για την 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 76. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική 13. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 79. Α, για μια στιγμή λέει η πρόεδρος. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη συμβιβαστική 13. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία γίνεται δεκτή με μία ψήφο διαφορά. 79 πρώτα, πρώτο τμήμα, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απερίφθη. 80. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 81. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 87. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 88. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. μπορεί να έχει απορριφθεί, αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 88 παρακαλώ ψηφίζετε. Πέραση ψηφοφορίας πράγματι απεριφθεί. «89 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 90 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 91 με προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Ποιοι είναι υπέρ. And but it's the same. Yeah, so the yeah. amendment was opposed yeah. the original. Thank you. Ε, that means that we vote on the original. Θα ψηφίσουμε μόνο το αρχικό λοιπόν κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. With um, the exact figures and the vote is open. Ψηφίζεται. It's already ε, Έγινε δεκτή με 30 ψήφους υπέρ. In favor, those... 93. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 96 κατά διέρεση ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτό το δεύτερο τμήμα, 97 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 98 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 99 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 100 ονομαστική, κατά ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή Το δεύτερο τμήμα της 104 τώρα ψηφίζουμε. Προσθήκη στην 12. Ονομαστική κλίση λοιπόν για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζεται το δεύτερο τμήμα της 104. Τέλος. Δεκτή. 24 υπέρ. 107. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος του δεύτερου τμήματος ψηφίζεται τέλος απερίφθη 108 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 109 υπέρ κατά αποχές Απερίφη. 111 Μα γιατί σηκώνονται, διαρωτάται η πρόεδρος. Κατάλαβα, είστε αρκετοί. Λοιπόν, ονομαστική κλίση για το πρώτο τμήμα της 111. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Α, και πάλι και εδώ είναι ονομαστική η κλίση, ψηφίζεται. Το δεύτερο τμήμα της 111. Τέλος της ψηφοφορίας. 37 υπέρ. 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 113 υπέρ. Α, δύο τμήματα πάλι ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το πρώτο κομμάτι ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ ξανά. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές δεκτό. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν του δευτέρου τμήματος της 113. Ψηφίζεται τέλος. Απερίφθη το δεύτερο τμήμα. 114. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι είναι αποχές, απερίφθη. 115. Υπέρ, κατά αποχές δεκτή 116 υπέρ κατά αποχές απερίφθεια. 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές απορρίπτεται Ας υπάρξει έλεγχος για την 120. Ψηφίζετε παρακαλώ. Τέλος. Ψηφίσατε όλοι. Απερίφθη. 121. με προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. 122 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφε. 123 ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. 124 ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απερίφε. 125 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 125, ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. 126 καταπίπτει, ψηφίζουμε την 127. Ποιοι είναι υπέρ. Εκατόν ψηφίζουμε, επαναλαμβάνει η πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ, ξανά. Κατά. Δεκτή η 127. 128. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές δεκτή. 129. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν απερίφη. 130. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Απερίφη. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απερίφη. 133 καταπίπτει, Τρία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Εκατόν τέσσερα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 135. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 4. Ψηφίζεται. Οι συντηρητικοί έχουν ένα επιπλέον. Απερίφθη. Με έξι ψήφους διαφορά ή τέσσερα. Περνάμε στην πέντε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Έξι. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν απερίφθη. Επτά. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Οκτώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Εννέα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Δέκα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Εντεκά υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 1 στις αιτιολογικές σκέψεις. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 15 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφη. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 25. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 26 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 27 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 31 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 32 και 33 μαζί υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 34. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πάντα ένας επιπλέον από τους συντηρητικούς. Εξακολουθεί να είναι ένας επιπλέον από τους συντηρητικούς. Πέρα της ψηφοφορίας Δεκτή. 27 ψήφοι υπέρ. Οπότε δεν έχει σημασία ακόμα κι αν ήταν ένας παραπάνω. 35 λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. 36 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε τώρα ονομαστική ψηφοφορία στην πρόταση νομοδότησης όπως τροπολογήθηκε. Τέλος. 34 υπέρ. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. for being part of the voting session now. Ωραία, ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Περνάμε στη συνέχεια της συνεδρίασής μας. Θα συζητήσουμε την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία. Οπότε θα έχουμε διερμηνία και στη νοηματική γλώσσα. Και επίσης έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες που θα βρείτε μπροστά σας. Αν ο μιλητής μιλάει πολύ γρήγορα και δεν κατανοείτε τι λέει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κίτρινη κάρτα. Αυτή είναι η πιο σημαντική. Δείχνει ότι ο μιλητής μιλάει πολύ γρήγορα. Για να περάσουμε στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης, λοιπόν.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 Okay, we are only five, six minutes. 5-6 λεπτά έχουμε μείνει πίσω, οπότε πολύ μικρή καθυστέρηση. Αλλά παρόλα αυτά ας περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα, που όπως σας προανέφερα είναι το σημείο 6 και αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνουμε και στην Επιτροπή μας όπως είπα και προηγουμένως, αν δεν παρακολουθείτε τη διερμηνία γιατί μιλάει πολύ γρήγορα ο μιλητής ή ομιλήτρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κίτρινη κάρτα. Αν έχετε πρόβλημα κατανόησης και δεν καταλαβαίνετε τι λέει ο μιλητής, μπορείτε να σηκώσετε την κόκκινη κάρτα για να το, το επισημάνουμε και να επαναλάβει με πιο απλά λόγια. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγητριά μας. Θα εξετάσουμε τις ε, πάνω από 400 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο έκθεση της κυρίας Χέλγα Στίβενς με θέμα την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην εισηγητριά μας, την κυρία Στίβενς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα θυμάστε ότι πριν από ένα χρόνο διοργάνωσα στο ημικύκλιο στην αίθουσα της Ολομέλειας ε, στις Βρυξέλλες μία διάσκεψη για να ε, γιορτάσουμε την πολυγλωσία και των νοηματικών γλωσσών που είναι μαζί με τις επίσημες 32. Ήταν πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία όπου και οι ομιλούμενες και οι νοηματικές γλώσσες ακούστηκαν στην αίθουσα στην οποία δούλευαν ταυτόχρονα τόσοι πολλοί διερμηνείς και ομιλουμένων γλωσσών και ε, νοηματικής γλώσσας. Ήταν πραγματικά ένα καταπληκτικό γεγονός, ένα φοβερό βίωμα, μια μοναδική εκδήλωση που μου δίνουν κουράγιο και ενέργεια. Είναι σημαντικές λοιπόν τέτοιες διοργανώσεις. Οπότε θα ήθελα με την έκθεσή μου να κάνω ένα βήμα ακόμη και να δώσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές κατευθυντήριες γραμμές και στόχους για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε και μετά το 2020 να εφαρμόζουμε τη στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία προκειμένου να υποφεληθούν όλοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας που έχουν κάποια αναπηρία στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες τώρα, με ιδιαίτερη, καταρχήν δίκαιο επισημανα, ε, επισημάνατε κυρία Πρόεδρε ότι έχουμε πάρα πολύ 300 τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που τις κατέθεσαν και να πω ότι ε, ε, χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί όλες οι τροπολογίες μου συνυπογράφησαν ε, και από πολλούς συναδέλφους ε, της Επιτροπής και από πολλά μέλη της διακομματικής ομάδας για τα άτομα με αναπηρίες. Και είμαι πεπισμένη ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τροπολογίες μου ε, εκπονήθηκαν μετά από στενή συνεργασία και πολλές διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις ε, ατόμων με αναπηρίες και έλαβα υπόψη όχι μόνο τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αναπηρία αλλά και των επιμέρους ονόσεων που εκπροσωπεί. Θέλω όλα τα άτομα με αναπηρίες να καλύπτονται από τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, εστιαζόμαστε κυρίως στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ώστε να δείξουμε την προστιθέμενη αξία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε αποτελέσματα. Ε, το πρόγραμμα Erasmus Συν θα πρέπει να συμμορφώνεται με το CRPD, την Σύμβαση για τα άτομα με Επίσης, έχουμε και το πρόγραμμα για την κάρτα αναπηρίας, που ελπίζουμε ότι θα ευδοκιμήσει και θα έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα με άλλες ευρωπαϊκές κάρτες. Σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, το σχέδιο συμβαστικών τροπολογιών ε, απεστάλλει χθε τους και οδησηγητές κατάφερα να συμπεριλάβω ένα ευρύ φάσμα τροπολογιών στις συμβαστικές, στις συμβαστικές μου τροπολογίες, ε, συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών και της Επιτροπής ε, Γυναικών. Βέβαια, δεν θέλω απλώ να αντιγράφουμε πιστά την έκθεση της περασμένης χρονιάς για την εφαρμογή ε, του CRPD, αλλά θέλω να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για μία απτή στρατηγική. Και για να το καταφέρουμε, σκοπεύω να διοργανώσω στην, στις εβδομάδες 41 ε, και 42 άλλες δύο συνεδριάσεις και εισηγητών και θα ήθελα να προετοιμάσω αυτές τις συνεδριάσεις, τις συνεδριάσεις ε, ε, και να τις επιταχύνουμε με προηγούμενη διαβούλευση με τους σκιώδεις ηγητές. Για να καταλήξουμε σε μία σύντομη αλλά περιεκτική έκθεση θα ήθελα να λάβετε υπόψη τις τροπολογίες των οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες, ώστε να καταλήξουμε σε διακομματικές τροπολογίες που θα τύχουν γενικές υποστήριξη. Πέρυσι, η έκθεσή μας για την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών ε, πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία και στην Επιτροπή Απασχόληση και στην Ολομέλη. Ελπίζω η ίδια επιτυχία να, επιτυχ... επαναληφθεί και φέτος, ώστε να επιδώσουμε μια χρήσιμη και στοχευμένη έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς όφελος όλων των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Και περιμένουμε ανυπομονησία τα σχόλιά σας και εδώ σήμερα και στις περαιτέρω συναντήσεις μας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Γεζοβιέτσκα, που εκπροσωπεί τον κύριο Πλούρα που αποουσιάζει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας διαβάσω τις απόψεις του κυρίου Μάρεκ Πλούρα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητή Χέλγα, με ενδιαφέρον διάβασα τις τροπολογίες που ήταν πολύ άριθμες. Το γεγονό ότι κατατέθηκαν πάνω από 400 τροπολογίες στην έκθεση δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον των συναδέλφων και τη σπουδαιότητα του θέματος ε, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία. Είμαι πεπισμένο ότι η πληθώρα των τροπολογιών θα εμπλουτίσει την έκθεση της ε, Helga Stevens, ε, επισημένοντα σημαντικά θέματα πολύ αναφερθήκαμε στη στρατηγική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδύλιων, ώστε σε συνδυασμό και με κρατικά και με ιδιωτικά κονδύλια να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη μόχλευση και να δώσουμε μια όθηση στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Επίσης, σημαντικό είναι ότι τονίζουμε πως τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να ε, στηρίξουν άλλες, άλλα Ινστιτούτα ε, και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε και τις απόμακρες κοινότητες ε, που δεν έχουν πρόσβαση. Επίσης, θέλουμε τις τροπολογίες να επιτρέψουμε την καλύτερη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, την αύξηση της προσβασιμότητας και την κατάργηση των φραγμών. Ε, πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για την παιδεία και την απασχόληση στις τροπολογίες τους και αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση αλλά και στην κατάρτιση και στην εργοπολιτική ε, απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά θα επιτρέψουν σε μια μεγάλη ομάδα των συμπολιτών μας να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και στο επίπεδο της μόρφωσης και στο επίπεδο της απασχόλησης. Θα πρέπει να αποφύγουμε κάποιες συστημικές παγίδες όπως είναι κάποιες ανελαστικότητες που υπάρχουν στο σύστημα και μια προθυμία ε, πρόσληψης ατόμων με αναπηρία. Πολύ σωστά επισημένα τα σημεία αυτά η κυρία Σδανόκα. Ε, περιμένω με ανυπομονησία τη συζήτηση για τις συμβαστικές τροπολογίες και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία προκειμένου να διαμορφώσουμε μια αξιόλογη έκθεση. Ευχαριστώ. Μάρεκ Πλούρα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπλινκεβιτσούτε απουσιάζει, αλλά θα την αντικαταστήσει η κυρία Ρε... Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, κολλείεται σήμερα η κυρία Μπλίνκεβιτσούτε. Μου ζήτησε όμως να, μεταφέρω, σας μεταφέρω το μήνυμά της. Θα ήθελα να πω ότι είναι η σκιώδη συγγήτρια σοσιαλιστών και δημοκρατών. Έχει καταθέσει 37 τροπολογίες στην έκθεση Στίβενς και οι περισσότερες αφορούν τα εξής θέματα. Καταρχήν, τη μνήμα των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων στην έκθεση, γιατί η κυρία Πλυνκεβιτσούτα θεωρεί ότι από πολλές απόψεις οι ηλικιωμένοι εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία. Του αφορά το θέμα. Επίσης, ζητά την συμπερίληψη μιας μνήας των προσωρινών αναπηριών. Και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές μιλούμε για ανθρώπου με λειτουργικούς περιορισμούς και που θα υποφελούνταν τα μάλα από την προσβασιμότητα. Θα πρέπει αυτή να εξασφαλίζεται για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η συμπερίληψη της μνήας στη σημασία που έχει η πρόληψη, τα μέτρα πρόληψης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και τη σημασία να παραμείνουν ενεργά τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Επίση, ε, απευθύνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνει τι ευρωπαϊκές προδιαγραφές προσβασιμότητα σε όλες τα δημόσια μέσα μεταφορά. Και κάτι πρακτικό και εύχριστο, η ανάγκη, ε, η, η κλίση, ε, η επίγουσα κλίση 112 θα πρέπει να είναι πλήρως προσιτή, αυτός ο αριθμός κλίσης 112 να είναι πλήρως προσιτό σε όλα τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης, ε, ζητά από το Συμβούλιο να ξεπεράσει το αδιέξοδο και να δρομολογήσει την οδηγία για την κατάργηση των διακρίσεων και επίσης επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία για το 2030 να περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να, να προωθούνται συστήματα κοινωνική προστασία χωρί αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα στα πλεονεκτήματα και τις υπηρεσίες των ατόμων με αναπηρίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ε, απευθύνεται έκλειστα κράτη-μέλη να θέσουν κάποια όρια κοινωνικής προστασίας για άτομα με αναπηρίες, ώστε να εξασφαλίζονται ε, να εξασφαλίζεται ε, αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Επίση, η ε, κυρία Πλυνκεβιτσούτε, θα ήθελα να ευχαριστήσει θερμότατα την εισηγήτρια την κυρία Στίβες για το πολύ αξιόλογο έργο της και προσβλέπει σε, σε μια αίσια διεκπαιρέωση των συζητήσεων και τη έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Σας ευχαριστώ και καταρχά. Όπω και σε άλλε περιστάσει ε, το έχω κάνει, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Έλγα Στίβεν για την πάρα πολύ εντελεχή δουλειά που έχει κάνει. Πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά για την έκθεση αυτή και ήμουν σε θέση να προσυπογράψω και να συνυπογράψω πολλέ από τι ε, τροπολογίε τη. Τι πιο πολλέ ε, είναι κάποιε για τι οποίε έχω κάποιε ερωτήσει. Κάποιε ερωτήσει που θα ήθελα να διευκρινιστούν. Για να αναφερθώ σε αυτά που είπε η Χέλγα και στην παρουσίασή της και στην παρέμβασή της, συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Erasmus. Θα πρέπει να είναι συμβατό με τη σύμβαση του για τα άτομα με αναπηρία και πιστεύω ότι η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να υποστηρίξει την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά τι συστάσει για την πράξη προσβασιμότητα, συμφωνώ επίση Να αναφέρω κάνα δύο πράγματα από τι δικέ μου τροπολογίε και ένα τελικό σχόλιο θα μου επιτρέψετε για τους συμβιβασμού. Για τις δικέ μου τροπολογίε θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει ανεξάρτητη ε, συνοδεία Είχαμε 300 άτομα χθε από 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια. Πάρα πολύ ισχυρό σαν μήνυμα, είτε στι Βρυξέλλε είτε στο Στρασβούργο. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και εμεί θα θέλαμε ως ομάδα η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων να ξεμπλοκάρει επιτέλου στο Συμβούλιο και να ακολουθήσουμε πιο έντονη διατύπωση από αυτή που προτείνει η συγκεκριτή. Έχουμε κάποιες τροπολογίες, αρκετές για το 883. Όπως ξέρετε το έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή μας το θέμα αυτό. Κάποια από αυτά τα στοιχεία λοιπόν μας βρίσκουν σύμφωνος, αλλά πιστεύω ότι παραπάνω κάπως. Είναι ενδεχομένως ε, όχι σωστή πρακτική να καθορίζει μία έκθεση τι δηλαδή θα μπει σε κάποια άλλη έκθεση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νομοθετική πρόταση. Αυτό συζητάμε ουσιαστικά στην Επιτροπή μα λίγο πολύ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την τροπολογία 883, ε, έτσι έχει διατύπωση, θα πρέπει να δούμε και τι πιστεύουν οι συνάδελφοι. και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες αυτές και γιατί κάποιες από τις τροπολογίες μιλάνε για τη λήψη αποφάσεων και τους α, τα άτομα, αναπληρωματικά άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις. Εδώ δεν έχω πραγματικά εμπειρία. Ούτε γνωρίζω το ζήτημα επακριβώς, αλλά μου φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αποχρώσεις. Αυτή η τοποθέτηση αυστηρή, άσπρο ή μαύρο μου φαίνεται ότι ενδεχομένω να μην ταιριάζει. Και είμαι εντελώ ανοιχτή και πρόθυμη να συζητήσω τι τροπολογίε αυτέ, να ακούσω τι έχουν να πούν και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί. Έχω όμω πολλέ απορίε ακόμα. Πέραν τούτου, δεν είχα χρόνο να εξετάσω τις συμβαστικές τροπολογίες αλλά δεδομένου το γεγονότος ότι έχω προσυπογράψει πολλές από τις τραπολογίες της ΕΛΚΑ, είναι βέβαια ότι θα καταφέρουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω το οτιδήποτε επακριβώς ε, σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία η κυρία Κούνεβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια η συνάδελφο Χαρίντα Στίβεν για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στην έκθεση για την αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική από την Αναπηρία. Με χαρά διαπιστώσα ότι έχει λάβει υπόψη τι όλε τι προτάσει των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία. Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος που επέλεξα να στηρίξω την προσπάθεια συνυπογράφοντας όλες τις τροπολογίες. Επιπλέον όμως θέλησα να αναδείξω ορισμένα θέματα που κατά τη δική μου γνώμη θα έπρεπε να υπογραμμιστούν στην στρατηγική. Και επιλέγω να αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα για να μπορέσω να συμβάλλω στην συζήτηση μας τη σημασία των δραστηριοτήτων αναψυχής ως μέσο ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία. Την ανάγκη ανταλλαγής καλών πρακτικών που αφορούν την ανεξάρτητη διαβίωση, ένα μοντέλο που ακόμα και στις πιο προοδευτικές χώρες βρίσκει προβλήματα εφαρμογής σήμερα. Την εξασφάλιση προσβασιμότητας των προϊόντων πολιτισμού και των υπηρεσιών τουρισμού. Την ενίσχυση των μέτρων θετικής διακρίση με την υιοθέτηση ελάχιστων ποσοστών πρόσληψης που τα αφορούν άτομα με αναπηρία. Αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε τα μέτρα λιτότητας να μην επιδρούν στο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μέτρα αντίσχυσης της ισότητας ατόμων που κινδυνεύουν από πολλαπλές διακρίσεις συμπεριλαμβανομένων και των ΛΟΑΤΚΙ με αναπηρία. Διοργάνωση εκστρατιών, ευαισθητοποίηση του κοινού, προστασία των αναπαραγωγικών και σεξουαλικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και καταπόλεμηση των σχετικών βίαιων και αναγκαστικών πρακτικών. Αυτά είναι τα βασικά σημεία των τροπολογιών που κατέθεσα στην έκθεση. Και πάλι θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει από την εισηγήτρια είναι παραδειγματική. Οφείλω να σημειώσω ότι τα πράγματα, το πρόγραμμα εργασίας του φακέλου είναι εντατικό και αυτό είναι ευτυχέ. Ελπίζω όλοι να εργαστούμε προς την ίδια κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες σε ένα τέτοιο θέμα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και το λόγο έχει η κυρία Στάνοκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να υποστηρίξω την προηγούμενη ομιλία την κυρία Κωνσταντίνκα, τη φίλη μου, σε ό,τι αφορά αυτό που ανέφερε για τι αντιφάσει. Χρειάζεται ομοφωνία σε ό,τι αφορά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βελτιωθεί. Προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη προσβασιμότητα στα άτομα με, τέτοιες, ε, με τέτοιους περιορισμούς. Αυτό που χρειάζεται δηλαδή για να συμμετέχουν σωστά στην κοινωνία. Και επίσης έχουμε πολλές τροπολογίες και πατριότητά μας στο σημείο αυτό είναι η απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινωνική προστασία και υγεία. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Στίβεντσα για τη δουλειά που έχει κάνει για να μπουν όλες τι τροπολογίες σε συμβιβαστικέ προτάσεις, φυσικά δεδομένες και της, ε, της έλλειψης χρόνου. Η... Ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για να κοιτάξουμε τις τροπολογίες δεν ήταν αρκετός για να μπορούμε να τις εκτιμήσουμε σε βάθος. Αλλά θα έχουμε και τις συναντήσει συναντήσεις των σκιωτών. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να είναι καλή τελικά η έκθεση και να καταλήξουμε σε συμβιβασμό για όλα. Σας ευχαριστώ λοιπόν κυρία Στίβεντς και πάλι. Ευχαριστώ Λεκή Πρόεδρος. Η κυρία Γκέα από το Διευθυντή δεν είναι παρούσα. Δεν την αντικαθιστά και κανένας. Ζουέλ μέλλα από το ΙΕΝΕΦ την οποία και εκπροσωπεί κρυσματά. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρου ε, τη κυρία Μελά. Μάλιστα λέει η πρόεδρο. Τώρα, αυτοί που έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Σπρίνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και σύντομος. και θα μιλήσω στα βουλγαρικά για το θέμα αυτό, μου επιτρέπετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν, Πρόεδρε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αδιαμφισβήτητο ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και αποτελεί και στόχο προτεραιότητας για μας η εξέβρεση της καλύτερης δυνατής διατύπωσης για την έκθεση αυτή είναι κάτι που μας απασχολεί. Και εξίσου κέρια σημασία είναι να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τα εντύπωτα χαρακτηριστικά όλων των κριτών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω αυτά που μας είπε και η κυρία Στίβενς ε, εισαγωγικά διάσκεψη λοιπόν που έλαβε χώρα το πρώτο ήμιση του έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να επιβεβαιώσω τις συνέπειες της διάσκεψης αυτής σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση. Την ευαισθητοποίηση για τις κατηγορηματικές ενέργειε που χρειάζονται. Χρειάζονται για να εφαρμοστεί πραγματικά αυτή η στρατηγική. Έχουμε δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου δεν υπάρχει καν νομοθεσία για την εφαρμογή της νοηματικής γλώσσας. Σε μία από τις δύο χώρες αυτές, μάλλον μία από τις χώρες αυτές είναι η Βουλγαρία. Η διάσκεψη λοιπόν Στην διάσκεψη αυτή υπήρξε λοιπόν μια ομάδα ατόμων από την Βουλγαρία που χρησιμοποίησαν την νοηματική. Όταν λοιπόν τα άτομα αυτά επέστρεψαν στη Βουλγαρία, καταρτίστηκε ένα νομοσχέδιο. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εκείνης ήρθα σε επαφή με την κυρία Στίβενς. Την ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου, γιατί μας βοήθησε ιδιαιτέρως βοήθησε και τους συναδέλφους μας. Μας παρέχει συμβουλές και πολύ πολύ πλούσιο υλικό για το ζήτημα αυτό. Δυστυχώς. Η ψηφοφορία στην Βουλγαρική Βουλή δεν στέφτηκε με ανάλογη επιτυχία. Ακούσαμε επιχειρήματα τα οποία παρεμποδίζουν την γοργή εφαρμογή και έγκριση του νομοσχεδίου. Η πλειοψηφία δεν υποστηρίξει τελικά το νομοσχέδιο. Διαρωτώ με όμως. Δεν θα ήταν απαραίτητο μετά από την έγκριση της δικής μας της έκθεσης. Δεν θα ήταν ώρα να αναλογιστούμε και ιδιαίτερες δράσεις εφαρμογής στα κράτη-μέλη τέτοιων μέτρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Και ενδεχομένω αν υπάρχει ανάγκη να εξετάσουμε το ενδεχόμενο νέα νομοθεσία, όπου υπάρχει νομοθεσία στα κρατημέλη ενδεχομένω να επανελεχθεί και να προσαρμοστεί η νομοθεσία αυτή. Θα ήθελα άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για όλη την υποστήριξη την οποία έλαβα από την κυρία Στίβενς για τη δουλειά που έχει κάνει για την έκθεση αυτή και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μια πολύ καλή αξιόλογη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λακή Πρόεδρο. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μα είπατε. Ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που δεν το λόγο. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ την κυρία Στίβενς γιατί όντως ε, πρόκειται για πάρα πολύ καλή προσπάθεια και όντως και σε διάφορες άλλες περιστάσεις έχουμε αναφέρει το πόσο σημαντικό είναι να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών για το θέμα αυτό. Αλλά αυτό ξέρετε ξέρετε μόνο από εμάς, από εμά και μόνο το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες και φυσικά δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουν προσυπογράψει πολλοί συνάδελφοι και εγώ έχω προσυπογράψει πολλά κομμάτια μαζί με άλλους συναδέλφους. Το κάθε αυτό το κείμενο θα είναι πραγματικά πρωτοποριακό. Υπάρχουν δύο στοιχεία λοιπόν που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό που είναι καταρχάς πολύ σημαντικό είναι να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα ασκεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ασκεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να το επεξεργαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ω τώρα, για να πούμε την αλήθεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το έχει κάνει αυτό με όλη της την καρδιά. Έχει σημειώσει κάποιες πρόοδους, δεν είναι τόσο δυναμική από θα έπρεπε όμως. Αυτό αφανώς. Κατά δεύτερον, Είχαμε ήδη κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, κάποια σχέδια τα οποία ήταν θετικά και πολύ έτσι, πρωτοποριακά. Ακριβώς λοιπόν για το λόγο αυτό. Και εμείς, αλλά και η Επιτροπή θα πρέπει να κινηθεί με πρωτοποριακό τρόπο. Πρόκειται για ένα τομέα όπου με τα μέτρα αυτά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την ανεξάρτηση διαβίωση των ανθρώπων αυτών. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, από τα ίδια μέσα, προώθησε ένα θετικό πρόγραμμα το 2013. Το έργο, λοιπόν, αυτό ήταν μια επιγραμμική νοηματική γλώσσα στο διαδίκτυο για δερμηνείς. 750.000 ευρώ. Σκοπός ήταν λοιπόν τα ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστούν προσβάσιμα για άτομα με αναπηρίες σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι την... Μετά την ολοκλήρωση όμως του προγράμματος αυτού, κάναμε μήπως τίποτε. Όχι, τίποτα. Τελική παύλα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν στο 2017. Άτομα με ακουστική αναπηρία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εμά ε, τους ε, βουλευτές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διάφορες δικαιολογίε μας λέει ότι, α, κοιτάξτε, χρειάζονται αναλύσεις, αυτό είναι το θέμα και το καθεξής. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι όμως στην Ευρώπη δεν μπορούν να έχουν πριν από τι εκλογέ τις καμία επαφή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό είναι πραγματικά παράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σα ζητήσω την υποστήριξή σας για τη δράση αυτή, την ενέργεια αυτή. Το τρίτο σημείο που ήθελα να δείξω είναι το εξή. Η σύνδεση μεταξύ στρατηγικής και εφαρμογής. Ευτυχώ το πακέτο προσβασιμότητας και κατάργησης των εμποδίων έχει προχωρήσει καλά. Και σε ό,τι αφορά τις λοιπές στρατηγικές στην Ευρώπη, θα πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση και περιμένουμε το συντομότερο δυνατόν απάντηση από πλευρά του Συμβουλίου τώρα. Thank you. Σας ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν τώρα στον επόμενο ομιλητή. Η κυρία, κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμότατα την Χέλγα ε, Στίβενς για την αγαστή συνεργασία που έχουμε και θεωρώ ότι η τελική έκθεση θα συμβάλλει τα μάλα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναπηρία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημεία. Τα επισήμανε και ο Μάρεκ Πλούρα. Πολύ σημαντικό είναι να διαμορφώσουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο ε, αρρωγής για τα άτομα με αναπηρίες ώστε να ζουν όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται στις τοπικές τους κοινότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να αποκτήσουν πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία οι άνθρωποι με αναπηρία. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να προωθούμε τα ταλέντα των ατόμων με αναπηρία, ώστε να κατανικήσουμε τους φόβους στην απροθυμία των εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες. Βέβαια, δεν ανάγκη αυτό να ασχολείται ε, μια ένωση αναπήρων για το θέμα αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία και τον τρόπο σκέψης των κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη. Γιατί για τις κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι τιμή και καμάρι να προωθούν και να αναδεικνύουν τα ταλέντα των ατόμων με αναπηρία. Ε, επίσης μπορεί κάποια σημεία να είναι αμφιλεγόμενα και να προκαλέσουν συζήτηση στο μέλλον, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι εμένα δεν μου αρέσει η η λέξη ανάπηρος. Όλοι σε κάποιο βαθμό είμαστε ανάπηροι. Και πολλές φορές ανθρώπους που χαρακτηρίζουμε ανάπηρους είναι άνθρωποι με πολλά ταλέντα. Και μάλιστα καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι ανάπηροι χρειάζονται να υπερνικήσουν χιλιάδες ε, εμπόδια που δεν τα αντιμετωπίζουν οι μη ανάπηροι αρτιμελείς και ειδικά ε, τα άτομα με αναπηρίες έχουν πολλές φορές πολύ ιδιαίτερα ταλέντα. Ευχαριστώ. Οπότε να ρωτήσω την κυρία Εμμανουέλ Γκράντς που είναι τη ματάρχησα ή μάλλον η κυρία Ημακουλάδα Πλασέσια έχει έρθει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κάποια σύντομα σχόλια από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επενέσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της. Για την έκθεση την οποία προετοίμασε και για το ότι συμπεριέλαβε ορισμένες τροπολογίες οι οποίες διευκρινίζουν κάποια από τα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής. Σας ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις σας λοιπόν. Νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές υπογραμμίζουν πολλούς τομείς οι οποίες είναι τομείς που ανησυχούν την Επιτροπή στα πλαίσια της εφαρμογής της στρατηγικής. Το θέμα της ποιότητας των μέτρων αυτών είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν εφαρμόζουμε τις διάφορες δράσεις. Το θέμα της προσβασιμότητας θα πρέπει να γίνουν βήματα σε σχέση με τη βελτίωση της πράξης για την, για την προσβασιμότητα. Υπάρχουν ε, βέβαια στον τομέα της απασχόλησης, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, δυσκολίες. Οι προτάσεις της έκθεσης είναι θετικές και συνιστούν ουσιαστικά καινοτόμα στοιχεία που θα βοηθήσουν να εφαρμοστεί η νέα στρατηγική. Να υπογραμμίσω επίσης ότι εξακολουθούμε την προσπάθεια του mainstreaming στον τομέα της προσβασιμότητας και κάποιες από τις προτάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Το ότι δεν αναφέρονται ονομαστικά στη παρουσίαση της στρατηγικής δεν σημαίνει ότι τις αγνοούμε και το θέμα της προσβασιμότητας και το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων και οι ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται στη βελτίωση της συλλογής στοιχείων, όπως επίσης και της χρήσης των κοινοτικών ταμείων, έτσι ώστε να μην αποκλείουν αυτούς οι οποίοι έχουν κάποια ε, τέτοιου είδους θέματα. Σχετικά με τις τροπολογίες για τις μελλοντικές πολιτικές, προφανώς θα τα υπόψη μας για τις προτάσεις που θα κάνουμε στο μέλλον. και στα πλαίσια της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής όλα τα στοιχεία τα οποία προτείνεται θα ληφθούν υπόψη. Περιμένουμε λοιπόν την τελική έκθεση, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την παρούσα συζήτηση και θέλουμε πάντα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας διευκρινίζοντας τις απορίες σας. Ίσως ε, να κλείσει τη συζήτηση η κυρία Στίβενς πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ και τους Σκιώδης και τους άλλους συναδέλφους για τα σχόλιά τους, για τα συγχαρητήριά τους. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε την βέλτιστη δυνατή έκθεση. Η δουλειά μπροστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πριν δύο εβδομάδες, στα πλαίσια της εξέτασης της πράξης για την προσβασιμότητα, πώς να το πω, ε, ε, υπήρξαν ορισμένες παρανοήσεις, για να το πω διπλωματικά, ε, για τις επιπτώσεις των εμποδίων αυτών στην κοινωνία, η ένταξη στην κοινωνία των ανθρώπων αυτών ε, γίνεται δύσκολη λόγω ακριβώς αυτών των εμποδίων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον σωστό δρόμο. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ενημερώσουμε το Συμβούλιο και να καταλάβει το Συμβούλιο πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι με αναπηρίες να ενταχθούν σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητας. Όταν συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες διαπιστώνουμε ότι σε πολλούς τομείς στον τομέα της προσβασιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ανθρώπων με αναπηρία είμαστε πάρα πολύ πίσω. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένα επιπλέον αποφασιστικό βήμα το οποίο να βοηθήσει να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την συνεργασία μας μαζί σας, θα διευκρινίσουμε ελπίζω τις απορίες οι οποίες υπάρχουν, οι προτάσεις που ακούστηκαν οι περισσότερες με βρίσκουν σύμφωνοι και θα συνεχίσω την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου και θα φτάσουμε ελπίζω στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο του 2017. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως, κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την λεγόμενη e-card, ηλεκτρονική κάρτα ε, κοινωνικών υπηρεσιών. Η κυρία Χάκεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κανονιστικά εμπόδια είναι από τα κύρια εμπόδια για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, υπάρχει η πεποίθηση ότι εξακολουθεί να υφίσταται τεράστιο δυναμικό για την ανάπτυξη και την απασχόληση, επιτρέποντας την πιο αποτελεσματική πρόσβαση σε εκείνου που επιθυμούν να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι με την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας έχει το δυναμικό να συμβάλλει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την αγορά, απλουστεύοντας τις διοικητικές διαδικασίες και επίσης ε, θεωρεί ότι θα απλουστευτούν οι διατάξεις περί ασφάλισης και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό πάντως η ηλεκτρονική αυτή οδηγία για τις υπηρεσίες ε, ε, να καλύψει μια σειρά κλάδων φοροτεχνικούς, ε, συμβούλους, λογιστικούς και τον κατασκευαστικό κλάδο και κάποιους άλλους τομείς όπως τα ταξιδετικά πρακτορία. Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι η πρόταση αυτή δεν θα χορηγεί επιπλέον δικαιώματα στους παρόχους υπηρεσιών. Ε, δικαιώματα που εξασφαλίζονται ήδη για αυτούς από την οδική και τις υπηρεσίες. Αυτά λέει σε γενικέ γραμμές η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι πολλά σημεία θα πρέπει να τα αναλύσουμε πολύ πιο διεξοδικά. Καταρχήν ένα γενικό σχόλιο. Κάποιοι κλάδοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτάχθηκαν ε, στις προτάσεις της οδηγίας για την ηλεκτρονική κάρτα διασυνοριακών υπηρεσιών και τα συνδικάτα αλλά και οι οργανώσεις εργοδοτών στον ίδιο κλάδο ήταν κατά της ε, πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν έχουμε λοιπόν τέτοια ε, μεγάλη διαμαρτυρία θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε αυτά που προτείνονται. Επίσης, ε, κάποια κοινοβούλια, για παράδειγμα το, η Γερμανική Βουλή, Bundestag, και η Αυστριακή Βουλή, ε, εξέφερα γνωμοδοτήσεις επισημένοντας την αντίθεσή τους με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε κάποια στιγμή εκλήθη, να λάβω μια απόφαση. Τι να κάνω. Να συνεχίσω την ανάλυση προσπαθώντας να βελτιώσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να υποχωρήσω και να πω όχι, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα ή πολλά σημεία που ενδεχομένως δημιουργήσουν πρόβλημα, οπότε σταματώ. Τελικά προσπάθησα να διερευνήσω αν υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροπολογιών που θα περιορίσουν την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για παράδειγμα Πρώτη, να αφαιρέσουμε τον κατασκευαστικό κλάδο από το πεδίο εφαρμογή της οδηγία και να περιορίσουμε αισθητά κάποιες εφαρμογές της ηλεκτρονικής κάρτας, στι ασφαλίσει κυρίως, για να δούμε αν μια πιο ε, συνοπτική πρόταση και πιο περιορισμένη και στα θέματα των προθεσμιών είναι ικανή να βελτιώσει αρκετά την πρόταση ώστε να γίνει αποδεκτή τελικά. Και αυτές τις προτάσεις ε, τις ε, περιέλαβα σε τροπολογίες που κατέθεσα. Για το σημείο αυτό η Bundestag έχει υποβάλει πολλά σχόλια, μεταξύ άλλων και για τη νομική βάση, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό, γιατί εμείς μόνο γνωμοδότηση ε, συντάσσουμε. Κατ' ουσία αρμόδια είναι άλλη επιτροπή. Πάντως, ε, κάτι που βρήκα ιδιαίτερα εύστοχο είναι ότι η πρόταση αυτή θα αντέστρεφε τη σχέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών, σχέσεις που κατα... κατοχυρώνονται στις συνθήκες, γιατί με βάση τις συνθήκες ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να ξεκινήσουν, προ... η Επιτροπή μπορεί να ε, ξεκινήσει προκατακτική διαδικασία αν, παρα... αν διαπιστώσει παραβίαση των συνθήκων ενώπιο του ΔΕΚ. Με βάση όμως την προτινόμενη οδηγία και τον κανονισμό που συμβαδίζουν, απαιτείται από τα κράτη-μέλη να αντιστρέψουν οποιαδήποτε αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΔΕΚ, να προσφύγουν δηλαδή στο ΔΕΚ πρώτα και να καταρρύψουν την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμά τους για παραγωγή νομοθεσίας. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό και αντιστρέφει την ισορροπία δυνάμεων ε, κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και ε, ακούστηκε η μορφή ότι η πρόταση αυτή επαναφέρει την αρχή της χώρας προέλευσης. Επίσης, δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ στις δικές μου τροπολογίες επιχείρησα να καλύψω κάποια από τα θέματα που σας ανέφερα, όχι όλα βέβαια, αλλά περιμένω με ενδιαφέρον τα σχόλια των συναδέλφων και θα δευτερολογήσω για να απαντήσω στις παρατηρήσεις τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν για την εισαγωγή. Από το ΕΛΚ, ο κύριος Σούσας θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τον σκιώδη εισηγητή μα από το ΕΛΚ, ο οποίος δυστυχώ δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία την κυρία Χάρκιν για την καλή δουλειά που έχει ήδη κάνει. Επί της αρχής ε, καλωσορίζω τον απότερο στόχο για την ε, επάνθυνση της ενιαίας αγοράς και να απλοποιηθούν οι διασυνοριακές δραστηριότητε. Παρ' όλα αυτά δεν επιτρέπεται στην διαδικασία αυτή να χάσουμε τα πρότυπα ποιότητας. Γι' αυτό λοιπόν έγινε πρόταση από πλευράς μας για την θεωρώ ότι είναι πολύ μάλλον κρίσιμη αυτή η πρόταση για την Ευρωπαϊκή αυτή ηλεκτρονική κάρτα για τι κοινωνικέ υπηρεσίε. Δεν έχει ακόμα ρημάσει, θεωρώ, επαρκώ η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει πάρα πολλέ αδυναμίε, ε, τι οποίε σίγουρα θα πρέπει να διορθώσουμε. Και όλο ιδιαίτερο θα πρέπει να φροντίσουμε να μην δημιουργηθούν παράλληλε δομέ. Θα πρέπει να κατανοήσουμε το ήδη υφιστάμενο ευρωπαϊκό επαγγελματικό πιστοποιητικό. Και επίση αναρωτιέμαι κατά πόσον πραγματικά είναι απαραίτητο να υπάρξει μια νέα υπηρεσία για τον συντονισμό, μήπω θα έχει νόημα καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε ήδη φυστάμενε δομέ. Κάτι άλλο που είναι απολύτω απαραίτητο. Τα κράτη-μέλη να έχουν και να λάβουμε υπόψη τι ε, αρμοδιότητες τους και τι εξισοδοτήσεις του. Ε, στη Γερμανία έχουμε ομοσπονδιακή δομή. Δεν τον υπεύθυνε, λοιπόν η κεντρική κυβέρνηση, αλλά τα μονομένα κρατήδια για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών. Αυτό δημιουργεί ακόμα πιο πολλά προβλήματα. Θα καταθέσω σχετικέ τροπολογίε και προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία με την εισηγήτρια, καθώ και με όλου του σκιώδει συζητητέ. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ, κύριε Ρέγκνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα αυτή εξ αρχή ε, να πω το εξή, ότι εδώ δεν έχουμε μια νομοθετική πρόταση όπω είναι πολλέ άλλε. Ε, εδώ πρόκειται για πολύ θεμελιώδει επεξεγήσεις και θέματα που έχουν πολύ βασική, βασικές και σημαντικέ επιπτώσεις σε όλους. Ε, φυσικά όλοι θέλουν να λειτουργεί η ενιαία αγορά, αλλά η ενιαία αγορά μπορεί να λειτουργεί μόνο κατά πόσον αυτοί που παρέχουν ε, υπηρεσίες μπορούν πραγματικά να προστατευτούν. Και γι' αυτό λοιπόν ήθελα να πω ότι η εσωτερική αγορά σκοπό έχει να εξυπηρετεί τελικά τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτός σκοπός. Στην πρόταση που έχουμε λοιπόν επί του επιτάπητος αυτή τη στιγμή δεν πιστεύουμε ότι αυτή η προστιθέμενη αξία αμφισβητείται έχουμε και την οδηγία για την παροχή υπηρεσιών, όπου εξακολουθούν να έχουμε πάρα πολλά ε, ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τους ομολόγους, για παράδειγμα, στις άλλες χώρες. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν, ξέρετε, εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια. Θα έπρεπε να τα διευκρινίσουμε πρώτα, κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την απόσπαση. Αυτό δεν μπορεί να διαχωριστεί από την χάρτα ε, υπηρεσιών εδώ η κατάσταση είναι η εξή Και οι υπηρεσίε και οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ευρώπη στον ορισμό των ατόμων που εργάζονται σε άλλα κρατημέλη θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον όντω πρόκειται για άτομο που παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες ή κατά πόσον πρόκειται για ψευδοαπασχολούμενο. Δεν αρκεί λοιπόν να τα καλύπτουμε όλα αυτά στην υπηρεσία για τους αποσπασμένους και μετά με την ε, χάρτα των υπηρεσιών να μην ρυθμίζονται αντίστοιχα τα πράγματα. Θα πρέπει να το δούμε όλο αυτό συνολικά στις μεμονωμένες τώρα διτάξεις ε, του κανονισμού. Να πω ότι η συγγήτρια έκανε και εισήγαγε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά θα κάνω, θέλω κάποιες ε, διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη διαγραφή ρητρών για τον τομέα της ασφάλειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πρόκειται για ουσιώδη ζητήματα όταν μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται διασυνοριακά. Όλοι λοιπόν στην αγορά θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τι υπηρεσίε, ε, τι ποιότητα έχουν οι υπηρεσίε αυτέ και ανάλογα θα πρέπει να λειτουργούν όλα αυτά λοιπόν. Και είμαι και μιλώ γενικά, αλλά η λειτουργία συμπεριλαμβάνει και ένα κάποιο έλεγχο ε, για να τηρούνται όλα αυτά ακριβώ. γιατί δεν έχει νόημα να υπάρχουν, για παράδειγμα, περιορισμοί στη ταχύτητα στου αυτοκινητοδρόμου, αν δεν υπάρχει το μηχάνημα να τα ελέγχει, η αστυνομία και το καθεξής. Το ίδιο ισχύει ασφαλώ και για τι υπηρεσίε. Τι υπηρεσίε που καλύπτονται από τη χάρτα αυτή και μπορούν να παρέχονται διασυνοριακά. Όλες οι πληροφορίε που έχω λοιπόν για του υπεύθυνου επιβολή των εθνικών αυτών νομοθεσιών διαπιστώνουν ότι δεν, υφιστα... δεν αρκούν οι υφιστάμενοι έλεγχοι. Αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετεί επαρκώ τα δικαιώματα το, της Ευρώπης. Για να υπάρχουν διασυνοριακές τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι και καλής ποιότητος για τον καταναλωτή, για τον εργαζόμενο, αλλά και για αυτόν που πραγματικά θέλει δίκαιο και θεμητό ανταγωνισμό για την αρχή της χώρας προέλευσης. Ουσιαστικά αυτό επανεισαγάγεται από την πίσω πόρτα. Οι ψευδοπασχολούμενοι πάλι Και αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι τομεί. Έχουμε αλλά ξέρετε δεν το συνηθίζω κιόλα. Έχουμε τομεί ε, οι οποίοι απαριθμούνται. Και ξέρουμε ότι στο θέμα της απόσπασης οι τομείς αυτοί μας προκάλεσαν και μας προκαλούν τεράστιες δυσκολίες. Και τώρα λοιπόν εδώ όλους τους βουλευτές θα ήθελα να τους ενημερώσω το σύστημα αυτό στην ε, θεωρία ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και φιλόδοξο να υπάρχει μια μεγενής ε, αγορά, αλλά θα πρέπει να τα εξετάσουμε τα συστήματα με πολύ ρεαλιστικό τρόπο, προκειμένου να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Να μην ξεκινήσουμε δηλαδή μόνο με τον κανονισμό, μετά με την οδηγία και μετά να συζητήσουμε τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο και αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αναπόσπαστο. Ω σύνολο λοιπόν θα πρέπει να το εξετάσουμε. Στην παρούσα λοιπόν φάση Αν ρωτιέμαι πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή υπεραξία. Εγώ προσωπικά δεν τη βλέπω και άρα το μόνο που έχω να συστήσω είναι να απορρίψουμε και να επικρίνουμε το σχέδιο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ε, ο Ρίρικε Τρεμπέζιος αποσιάζει κάποιος που την αντικαθιστά από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Όχι. Πάμε στην ΚΟΕ. Αλλά δεν βλέπω κανέναν ούτε από την ΚΟΕ. Η κυρία Ζητανοκά, από τους πράσινους παρακαλώ. Ε, είμαι ευγνώμων στη Μάριαν Χάρκιν και τους προλαλήσαντες που αμφισβήτησαν το δόκιμα της πρότασης. Και εμείς έχουμε πολλά ερωτηματικά και απορίες που προέκυψαν με την εξέταση της πρότασης. δεν είμαστε σε θέση προς το παρόν πάντως να, να κάνουμε μια θεωρητική, μια καλή αξιολόγηση της πρότασης. Σε ό,τι αφορά μια σωστή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματική Κάρτας, που είναι σχετικά πρόσφατη, τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2016, δεν πέρασαν ούτε δύο χρόνια. Γιατί δεν μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενημέρωση για το πώς έχει λειτουργήσει αυτή η κάρτα και μια αξιολόγηση σε σύγκριση και με τη νέα πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών. Βέβαια, η κάρτα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσφέρεται στους παρόχους υπηρεσιών ε, σε εθελούσια βάση. Αλλά από την πρόταση δεν προκύπτει κάτι τέτοιο με σαφήνεια. Ε, φοβόμαστε ότι θα επιβαρύνει περαιτέρω τους επιχειρηματίες και τους παρόχους υπηρεσιών. Κυρίως εκείνους που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε, στο κράτος υποδοχής ε, μόνο άπαξ ή προσωρινά προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Εκτιμώ λοιπόν ιδιαίτερος ε, την αναγκερθήσα βούληση της κυρίας Χάρκη να περιορίσει το πεδίο εφαρμογή της πρότασης της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο, εκτός βέβαια και αν ε, απορρίψουμε σε την πρόταση. Γιατί όπως σας είπα, έχουμε και εμείς πολλές αμφιβολίες και προβληματιζόμαστε τη, τι στάση να ακολουθήσουμε. Περιμένουμε πρώτα τις ε, συγκεκριμένες προτάσεις της εισηγήτριας και μετά θα λάβουμε θέση από αυτόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαχτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πρέπει να απλοποιήσουμε την διοικητική περιπλοκότητα. Ακούγεται σαν ε, μια καλή πρόταση. Σχετικά με την έκθεση αυτή, η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Υπηρεσιών στόχος είναι ε, διαφορετικός και αυτό για τρεις βασικούς λόγους. Και εδώ έρχομαι στις προηγούμενες παρεμβάσεις της κυρίας Χάρκιν ο πρώτος λόγος είναι ότι στόχος είναι η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της κατάργησης των εμποδίων στις διασυνοριακές συναλλαγές. Με άλλα λόγια, συνάδελφοι, το έγγραφο αυτό θέλει να περιορίσει τις αρμοδιότητες που έχουν τα κυρίαρχα κράτη που θα προσπαθούσαν να περιορίσουν τις παροχές υπηρεσιών στο έδαφος τους. Αυτό ήταν ο πρώτος λόγος. Βλέπουμε ότι πολλοί τομείς φοβούνται ότι αυτό το φαινόμενο θα ενταθεί, θα αυξηθεί ο αριθμός των ψευδοαυτοαπασχολούμενων και γι' αυτό ακριβώς η πρωτοβουλία της εισηγήτριας είναι μια καλή πρωτοβουλία γιατί θέλει να περιορίσει τα επαγγέλματα τα οποία θα μπορούσαν να εποφεληθούν αυτής της ηλεκτρονικής κάρτας. Και τρίτον, πιστεύουμε και νομίζω ότι περισσότεροι ανησυχούν ότι η κάρτα αυτή θα ενισχύσει το κοινωνικό dumping επιτρέποντας τους ξένους να μην εκπληρούν ορισμένες διαδικασίες αδειοδότησης και ορισμένα δηλωτικά διοικητικά τουλάχιστον σε ό,τι ισχύει στη Γαλλία. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί λοιπόν όπως και η κυρία Χάκιν. Ευχαριστώ πολύ η επόμενη ομιλήτρια. Θα ήθελα να αναφερθώ, Πρόεδρε, ε, στις υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να καλύπτονται από την ε, e-card. Πρόκειται για ένα εθελοντικό, θα έλεγα, μέσο είναι ένα πείραμα να το πω αλλιώς, μια απόπειρα καλύτερα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Είναι κάτι το οποίο αξίζει κανείς να διαπραγματευτεί και να συζητήσει. Θα πρέπει να δούμε όμως αν είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε ε, μέσω των τροπολογιών μας. και διευκρινίζει τα επαγγέλματα η κυρία Χάρκιν όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα αυτή. Εγώ έχω και κάποιες άλλες ιδέες. Πάντως, αν αρνηθούμε τη χρήση του μέσου αυτού, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους ε, ενίσχυσης, αν θέλετε, ή βοήθειας της ε, κινήσεις ε, και για τις συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε καλύτερη αναγνώριση των ικανοτήτων και των σπουδαστικών πιστοποιητικών. Δεν θα είναι κάτι το υποχρεωτικό. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν αν θα υιοθετήσουν ένα τέτοιο μέτρο. Νομίζω ότι μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Είναι κάτι το αποδεκτό για να υπάρξει καλύτερο συντονισμός υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και για να υπάρξει μια μορφή βελτίωσης όχι μόνο των εργοδοτών και των εργαζομένων αλλά και για την ποιότητα των υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Χάκινγκ. Μήπως ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Στράους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, γεια σας. Ε, δεν άκουσα το πρώτο κομμάτι της ε, παρέμβασης της κυρίας Χάρκινγκ, αλλά νομίζω ότι έχω καταλάβει την ουσία και άκουσα και τα σχόλια και τις προτάσεις ε, οι οποίες έχουν γίνει πάνω στην δική μας ε, πρόταση. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχει αρκετή ανησυχία γύρω από τις προτάσεις που έχουν γίνει για την e-card και κάποιες από αυτές τις ανησυχίες εκφράστηκαν και εδώ. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε πάρα πολύ δεκτικοί στους τρόπους βελτίωσης του συγκεκριμένου μέσου η οποία δεν κάνει βήματα επιπλέον της ισχύουσας οδηγίας, αλλά λέει ότι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν γίνει δεκτές από το σώμα σας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γίνουν πραγματικότητα. Το θέμα της αρχής προέλευσης έχει έλθει πολλές φορές εδώ και η πρόταση ε, δεν θίγει αυτή την βασική αρχή, παραμένει η αρμοδιότητα της κράτους χώρας προέλευσης η οποία πιστοποιεί ότι ο παροχέας της υπηρεσίας ε, λειτουργεί στο έδαφος της συγκεκριμένης χώρας. Κατά τα όλες οι εξουσίες, όλες οι αρμοδιότητες, όλοι οι έλεγχοι ρυθμιστικοί και διακανονιστικοί παραμένουν στα κράτη-μέλη. Δεν αλλάζουμε κάτι δηλαδή ως προς αυτό. Τώρα για τους τομείς τους οποίους η e θα μπορούσε να διευκολύνει κάποιες ψευδοεπιχειρήσεις ή κάποιους ψευδοαυτοαπασχολούμενους κτλ. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Μέσω της e-card θα είναι πολύ εύκολο για τη χώρα που φιλοξενεί την υπηρεσία να ελέγχει. Μπορεί οι επιχειρήσεις να μην ζητούν την e card είναι έτσι και αλλιώς κάτι το εθελοντικό, να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε μια χώρα άλλη της δικής τους με διαφορετικό τρόπο. Συνεπώς λοιπόν, στον βαθμό που θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα και στον βαθμό που τα κράτη-μέλη θέλουν να την χρησιμοποιήσουν για να διευκολύνουν τις μορφές ελέγχου, θα το κάνουν και θα μειώσει τις, α, ε, ε, ε, ευκαιρίες που υπάρχουν για την ύπαρξη εταιριών γραμματοκιβωτίων. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση ε, βοήθησε για να ε, διευκρινίσουμε τον προβληματισμό και την ανησυχία των συναδέλφων. Και ε, επισημάναμε ότι ό,τι προβλήματα προκύψουν από την οδηγία και τις υπηρεσίες θα μεγιστοποιηθούν με την εισαγωγή αυτής της πρότασης για τις ηλεκτρονικές ε, κάρτες για τις υπηρεσίες. Μερικοί κίνδυνοι είναι ορατοί και πραγματικοί και άλλοι είναι πιθανοί. Αλλά ε, υπάρχει προβληματισμό. Μπορεί να είμαστε πολύ απαιτητικοί, μπορεί να ζητούμε τον ουρανό μετάστρα. Θα πρέπει να το ξαναζητήσουμε με τους συναδέλφου. Πάντως η πρόταση αυτή έπρεπε ήδη να είχε ε, εντοπίσει και λύσει κάποια προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Προς το παρόν μόνο ερωτήσεις έχω, απαντήσεις δεν έχω βρει. Θα, θα διερευνήσω περαιτέρω πάντως όλα αυτά τα θέματα. Η κυρία Σόιντροβα είπε ότι είναι προαιρετικό το σύστημα. Ναι, είναι προαιρετικό για τις εταιρείε. Αν όμως οι εταιρείε αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές κάρτες μετά, είναι υποχρεωτικό για τις χώρες. Οπότε δεν μπορούμε απλώς να λέμε ότι είναι μόνο σε θελούσια βάση. Συμφωνώ με την άποψη ότι πρέπει να πούμε ε, η οδηγία αυτή υλοποιεί τους στόχους που αναγγέλει. Και συμφωνώ με τους συνάδελφους ε, ε, με το ΕΛΚΟ ότι υπάρχουν κάποια πρόβλα, προβλήματα με τις παράλληλες δομές, με τη σαφήνεια και με, την, ε, με το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης. και αυτά εντοπίστηκαν στο διατακτικό. Διαφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά του πιθανού κινδύνου να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές κάρτες από του ψευδοαπασχολουμένου. Δεν είναι απλώ ε, ε, φόβος, είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα που υπάρχει γιατί δεν δημιουργεί ασφάλεια δικαίου η διατύπωση της πρότασης και δημιουργεί ε, πρόσφορα για κατάχρηση οι εταιρείε και οι καταναλωτέ στα κράτη-μέλη υποδοχής οφείλουν να ε, εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες ανταγωνισμού με αυτού που έρχονται να προσφέρουν τι υπηρεσίε. Δεν μιλούμε δηλαδή μόνο για τι εταιρείε που παρέχουν υπηρεσίε διασυνοριακά. Μιλούμε για συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού και εντό των κρατών μελών. Και συμφωνώ με τον με το συνάδελφο από τους σοσιαλιστές ότι έχουν ε, απομείνει αναπάντητα ερωτήματα για την ποιότητα των υπηρεσιών, για παράδειγμα και για το, το θέμα της συμμόρφωσης ε, με τους κανόνες. Από ό,τι ξέρω ξανά τέθηκε μια προθεσμία. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και πολλές ε, συζητήσεις, πάντως προσβλέπω ε, στη συνεργασία με τους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Το χρονοδιάγραμμα που έχω εγώ τουλάχιστον προβλέπει προθεσμία για τις τροπολογίες την 24η Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι με εξέταση των τροπολογιών στις 9 Νοεμβρίου. Yes, uh, it's uh, the consideration of amendments table. Μάλλον 20 Νοεμβρίου θα γίνει εξέταση των τροπολογιών 20 Νοεμβρίου 2017 και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας αρχικά έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου και δεν ξέρουμε ακόμη σε ποια ολομέλεια θα γίνει η τελική ψηφοφορία. Ωραία, ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα. Περάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης την οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του του Κοινοβουλίου για το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ηλεκτρονικής, της ε, Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Κάρτας για τις υπηρεσίες. Αυτό, αυτή η πρόταση αποτελεί ένα τμήμα του νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου και αποτελεί αρμοδιότητα της κυρίας Σόιντροβα που είναι και συντάκτηρια της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αντικείμενο της συζήτησης είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης ε, για την Ευρωπαϊκή Ελεκτρονική Κάρτα για τις Υπηρεσίες. Ε, να υπενθυμίσω ότι είναι προαιρετική αυτή η ηλεκτρονική κάρτα και στόχο έχει να πλουστεύσει τα πράγματα και να άρει τους φραγμούς ε, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν σε διασυνοριακές ε, δραστηριότητες στον κατασκευαστικό τομέα. Και η πρόταση αυτή συνδέεται κάπως και με την οδηγία για τις υπηρεσίες και μάλιστα βελτιώνει την κατάσταση, αν και δεν αξιοποιεί στο έπακρο το δυναμικό αυτή η πρόταση. Περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών. Η προλαλή σα η τη της προηγούμενης η κυρία, η Χάρκιν, είπε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα σωστό εργαλείο για την εφαρμογή. Εμείς προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις για να επεκτείνουν τις τις δραστηριότητές τους και στα άλλα κρατημέλη. Γιατί μέχρι στιγμή δεν υπάρχει υποχρέωση για αυτές τις επιχειρήσεις. Αν υπήρχε η, μια τέτοια κάρτα υπηρεσιών υποχρεωτική, θα ήταν ε, υποχρεωτικό και για τα κράτη-μέλη να προσφέρουν υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και να τις διευκολύνουν να επεκταθούν. Θα υπήρχε δηλαδή υποχρέωση έκδοσης της ηλεκτρονικής κάρτας. και οι επιχειρήσεις θα ήταν υποχρεωμένες να παράσχουν πολλές πληροφορίες για να ξεκινήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλες χώρες. Οπότε η πρόταση αυτή κατά τη γνώμη μου έχει ένα πλεονέκτημα. σήμερα οι επιχειρήσεις μπορούν να αποταθούν σε επιμελητήρια, σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις της χώρας υποδοχής. Αλλά η χώρα υποδοχής δεν υποχρεούται να παράσχει αυτές τις πληροφορίες. Τώρα, όταν η επιχείρηση ζητά έκδοση κάρτας στη χώρα υποδοχής, το πλεονέκτημα που προσφέρει η πρόταση είναι ότι η επιχείρηση θα έχει άμεση επαφή με τις αρχές της χώρας υποδοχής, της χώρας προέλευσης μάλλον, και θα πρέπει να τηρεί όλε τι υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος στη χώρα προέλευσης και αυτό γίνεται, κοινοποιείται στη χώρα υποδοχής. Πάντως, ο κανονισμός δεν απλουστεύει πρότυπα ή προδιαγραφές που ισχύουν στα άλλα κράτη-μέλη. Δεν τα επηρεάζει. Αφορά μόνο μια διοικητική διαδικασία για τις επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνομαι τις αφιβολίες και τις ανησυχίες των συναδέλφων για κίνδυνο κατάχρησης της κάρτας αυτής. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να προβλέψουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες μέσω των τροπολογιών μας. Τώρα για να δούμε το κείμενο. Θα ήθελα να καταθέσω τροπολογίες που ήδη έχω και που εξασφαλίζουν αυτέ τι ασφαλιστικέ δικλείδε που σα ανέφερα. Θα πρέπει να τονίσουμε καταρχήν τον προαιρετικό χαρακτήρα τη ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών. Αυτό πρέπει να είναι σαφέ. Επίση, ε, η κάρτα θα πρέπει να ισχύει για 24 μήνες και να ανανεώνεται αυτομάτως για το ίδιο χρονικό διάστημα με την επιφύλαξη όμως ότι έχουν ε, ελεγχθεί τα στοιχεία και η εγκυρότητα των στοιχείων που αφορούν τον πάροχο υπηρεσιών. Έτσι, με τον έλεγχο της εγκυρότητας των στοιχείων που αφορούν τον πάροχο υπηρεσιών, εξασφαλίζουμε μία βεβαιότητα. Επίσης, για την πρακτική της σιωπηρής ε, συγκατάθεσης. Αυτό ίσχυε στο παρελθόν. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στην συγκεκριμένη κάρτα, γιατί όπως σας είπα είναι προαιρετική, σε εθελοντική βάση. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι η αρχή της σιωπηρής αποδοχής της κατάθεσης δεν είναι απαραίτητη. Και μια και οι δύο χώρες θέλουν μια βεβαιότητα, καλό θα είναι να υπάρχει κάποια, κάποιος έλεγχος. Οπότε διαγράφεται η δυνατότητα της σιωπηρής ε, συγκατάθεσης. Επίσης, προτείνεται ενημέρωση των στοιχείων, επικαιροποίηση και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών δεν υποβάλλει τα ενημερωμένα στοιχεία. Και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στο κείμενο, κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι οι σχετικές τροπολογίες θα, θα βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιμένω τα σχόλια της σχετικά. Πάντως, για τις τροπολογίες αυτές είχαμε διαβουλεύσεις και με συνδικάτα και με οργανώσεις εργοδοτών, με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων, γιατί ε, είχαν και οι κοινωνικοί εταίροι αρκετέ αμφιβολίες για την πρόταση. Πάντως, ε, θα συνεργαστώ και με τους σκιώδης ηγητές για να τελειοποιήσω το κείμενό μου. Η οδηγία καλό θα είναι να έχει την υποστήριξη των κρατών μελών, αλλιώς ε, δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ρίγνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την οδηγία έχω να πω τα ίδια για τα οποία, τα οποία έχει πάει για τον κανονισμό. Οι πιθανότητε ε, και τα φατικά είναι ενδεχομένω πολλά, αλλά είναι τόσο μεγάλη και κίνδυνη που προς το παρόν έχω να πω ότι κλείνω και δεν μπορώ παρά να συστήσω την απόρρευση της πρότασης αυτής και θα ήθελα να πω με σαφήνεια ότι εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που είπε η κυρία Σόιντροβα για τις απαραίτητες βελτιώσεις. Εκτιμώ ιδιαίτερως ότι τα κάνετε τη δουλειά αυτή. Ωστόσο δεν αρκεί αυτό. Γιατί είναι τεράστιοι οι κίνδυνοι που ενέχονται να δώσω δύο παραδείγματα για να σας πω πόσο περιπλοκή είναι η κατάσταση. Εδώ αναφέρονται ιδιαίτερως ε, και παραδοσιακά επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών διασυνοριακά. Να δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα που νομίζω που μιλάει από μόνο του. Στην, ε, στις οικοδομές. Στην Αυστρία, στις οικοδομές, ε, και αυτό φαντάζομαι ισχύει παντού, όταν γίνεται έλεγχος επιθεώρηση, διαπιστώνεται ότι μάλιστα εδώ πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, συσσαγωγικά, κλασικό συσσαγωγικά ειδικό. Κλασικό λοιπόν, κλασική ερμοδιότητα ενός ε, εργάτη στην Αυστρία και συχνά διαπιστώνεται ότι το άτομο αυτό απασχολείται ως αυτοαπασχολούμενος. Σε ελέγχους λοιπόν τελικά καταλήγουμε ότι σε ό,τι αφορά την οδηγία ο επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κλασικός επιχειρηματίας αλλά ουσιαστικά αποτελεί και πληρεί όλες τις προδιαγραφές για εργαζόμενος. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται και σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Και θα το αντιμετωπίζαμε σε ό,τι αφορά τη χάρτα για τι υπηρεσίες αυτέ. Πώ θα, πώς θα μπορούσαν λοιπόν οι αρχέ, να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα ψευδοαπασχολούμενα. Πώ θα μπορούσαν να τα ελέγξουν καν. Αρκούν τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μα στην αντιγεία. Κυρία Σόιντροβα, είπατε τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να καταλήξουμε σε μια τέτοια εύρυθμα λειτουργούσα ενιαία αγορά. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι όχι να ξεκινήσουμε με μια χάρτα παροχής υπηρεσιών, αλλά με μια ευρωπαϊκή συνεργασία των σχετικών αρχών. Πώς είναι δυνατόν όταν ένας πάροχος υπηρεσιών, ένας επιχειρηματίας, εγώ να πάω ως Αυστριακή στην Ισπανία, στην Εστονία, και αναφέρεται στα γερμανικά. Τι άδεια έχω και τι θα κάνουν δηλαδή οι αρχές στην Εστονία. Θα πρέπει να τα μεταφράσει ο καθένας στη γλώσσα του. Είναι τόσο λοιπόν τρατηματικά που ενέχονται στην πρόταση αυτή που δεν μας επιτρέπουν να συγκαταθέσουμε, να συνενέσουμε με, το, με την πρόταση αυτή. Όλοι θέλουμε να λειτουργεί η αγορά εργασία και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει πραγματική συνεργασία μεταξύ των ε, υπηρεσιών. Έχω εκατοντάδε ιστορίε τέτοιε να σα πω. Δεν θέλω να σα κάνω να παρατηρείτε. Δυστυχώ δεν λειτουργεί αυτό επαρκώς. Όταν έχουν τέτοιε ανταλλαγέ οι υπηρεσίε των διάφορων χωρών για το κατά πόσο πληρούνται οι σχετικοί όροι και κατά πόσο εφαρμόζονται η σχετική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα άτομα τα οποία θέλουν και σκοπεύουν να παρέχουν τέτοιε υπηρεσίε τελική ανάλυση. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν. Σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά που είχα να πω τα είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Ε, ευχαριστώ αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο εισηγητής, κάποιες ρήτρες προστασίας δηλαδή. Θα ήθελα να προχωρήσω περισσότερο από ό,τι το έκανε εκείνη να συμπεριλάβω και τον τομέα των οικοδομών, τον κατασκευαστικό τομέα. Ε, αναφέρεται στην κατάργηση της λεγόμενης έμεσης, ε, ε, έμεσης ή σιωπηλής συμφωνίας. But as I said, we, we need to look at this further. Uh, I just have a question. Για το θέμα της σιωπηρής συνένεσης ήταν προηγούμενη παρατήρηση. Ε, αν εκδοθεί μια e-card για αόριστη περίοδο μπορεί σε μια ιστερότερη φάση μια χώρα υποδοχής να καταθέσει αντιρρήσεις. Ή εμποδίζεται η συγκεκριμένη χώρα. Γιατί αποκλειστικά θα χρησιμοποιήσουν επιχειρήματα όταν δόθηκε η αρχική άδεια. Θέλω να πω αλλιώς την ερώτησή μου. Υπάρχουν περιορισμοί για τις χώρες που φιλοξενούν τις δραστηριότητες αυτές εφόσον έχουν εκδώσει στο παρελθόν την e-card και για κάποιο λόγο σε μια ιστερότερη φάση θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν θέση. Υπάρχουν λοιπόν δεσμεύσεις, περιορισμοί εκτός από αυτούς ε, που προβλέπονται από την οδηγία ε, για τις υπηρεσίες. Δηλαδή, να το πω ξανά, αν έπρεπε να θέσουν ορισμένα θέματα και δεν το έκαναν αυτό τη στιγμή που κατατέθηκε ε, το αίτημα, τότε σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Η κυρία Ρέγκνερ αναφέρθηκε και στα θέματα τα οποία μπορεί να ισχύουν σε μία χώρα και την e-card και αν αυτό ε, θα επηρεάσει άλλες χώρες που εκδίδουν ή μπορεί να εκδίδουν ή μπορεί να μην εκδίδουν ε, τις ηλεκτρονικές αυτές κάρτες. Ευχαριστώ κύριε Χάρκιν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαρτάν και μετά στην Επιτροπή για να κλείσει. Κύριε Μαρτάν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα διστακτικός σχετικά με την οδηγία αυτή για το νομικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Κάρτα Υπηρεσιών. Και βλέπω ότι δεν είμαστε οι μόνοι που είμαστε τόσο διστακτικοί και σκεπτικιστές. Αυτόματη ανανέωση και απεριόριστη ανανέωση, απλή δήλωση φαλκίδευσης της κάρτας αδυναμία των κρατών μελών να θέσουν νέες απαιτήσει, ακόμα και αν ε, η κάρτα δεν έχει ακόμα παραδοθεί. Νομίζω ότι το νομικό πλαίσιο το οποίο ε, προτείνεται ε, αποδεικνύει την τεράστια χαλαρότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στερεί την χώρα από τα δικαιώματα της. Τι γίνεται με ένα δικαίωμα αν αλλάξει ανάμεσα σε δύο ανανεώσεις η εθνική νομοθεσία. Τι γίνεται σε επίπεδο νομικό αν ένας παροχέας κατηγορηθεί επανειλημμένα για αφαλκίδευση των καρτών. Του αποσύρεται η κάρτα αυτή. Νομίζω ότι το νομικό πλαίσιο αυτό έχει πάρα πολλές ατέλειες και επαναλαμβανόμεθα συνεχώς εδώ, η επιθυμία μιας πιο απόλυτης ελεύθερης αγοράς οθεί τον Ευρωπαίο νομοθέτη να αγνοεί περιφρονητικά την α, κυριαρχία των κρατών μελών. Και γι' αυτό προφανώς η τροπολογίες μας θα ακολουθήσουν την αντίθετη κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Στράους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Χάρκιν μόνο γενικώ. Όχι, απαντήστε σε όλες. Θα απαντήσω τις ερωτήσεις της κυρίας Χάρκιν τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να διαφυλάσσουν όλες τις ε, εξουσίες τους για να διερευνήσουν και ενδεχομένω να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν την ηλεκτρονική κάρτα ενός παρόχου υπηρεσιών. Εφόσον υπάρχουν νόμιμοι βάσιμοι λόγοι ότι κάτι πάει στραβά, το γεγονός ότι έχει εκδοθεί μια ηλεκτρονική κάρτα που δεν είδε να στερεί από το κράτος μέλος τη δυνατότητα να κάνει έρευνες είτε με επιτόπιους ελέγχους και αν ε, εντοπίσει σταλίες, ε, να ανακαλέσει, να αναστείλει. Οπότε διατηρούνται τα δικαιώματα των κρατών μέλων. Τώρα, η ανάκληση της ηλεκτρονικής κάρτας σε ένα κράτος μέλος ε, έχει συνέπειες σε άλλες χώρες. Αν το πρόβλημα ανέκυψε στο, στη χώρα υποδοχής, ναι. Αν όμως το πρόβλημα υπάρχει στο, στη χώρα προέλευσης, αν ε, ε, παράνομα παρέχει υπηρεσίες ε, ο πάροχος, τότε η ανάκληση στο κράτος υποδοχής έχει συνέπειες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε από αυτήν την άποψη είναι πανευρωπαϊκή εφαρμογή της αναστολής, σε περίπτωση που το πρόβλημα ανακύπτει στο κράτος προέλευσης η ε, κυρία Ρέγνερ ε, επισήμανε κάποια προβλήματα που ανέκυψαν στην Αυστρία. Η ηλεκτρονική κάρτα, και σας κουράζω γιατί επαναλαμβάνομαι, πρέπει να διευκολύνει τη δυνατότητα ε, των κρατών μελών, των αρμόδιων αρχών να εντοπίσουν φαινόμενα ψευδοαπασχόλησης. Αν ο πάροχος υπηρεσιών είναι αυτοαπασχολούμενος στη χώρα προέλευσης, θα ήταν δύσκολο να λάβει τέτοια ηλεκτρονική κάρτα. Γιατί για να λάβει κάποιο ηλεκτρονική κάρτα και να είναι δικαιούχο τέτοια κάρτα, θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσία στην ε, χώρα προέλευση, στη χώρα καταγωγή. Όχι να είναι αυτοαπασχολούμενο. Οπότε, μια και πρέπει να περάσει τη διαδικασία, πρέπει να καταθέσει αποδείξει. Ε, σίγουρα ε, η Ευρωπαϊκή Κάρτα δεν διορθώνει μια κατάσταση που είναι ήδη καταχρηστική, αλλά ούτε διευκολύνει μια τέτοια κατάχρηση τη ψευδοαπασχόληση. Αντίθετα, η δυνατότητα που έχουν οι ε, αρμόδιες αρχές με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων είναι να ελέγξουν αν οι ισχυρισμοί του παρόχου υπηρεσιών είναι έγκυροι. Ευχαριστώ. Και τελευταία ομιλήτρια, η συγγετριά μας, η κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να πω ότι εγώ δεν είμαι υπέτεια για την ε, εκπόνηση της οδηγίας, εγώ είμαι απλώς συντάκτρια της γνωμοδότησης. Και καθήκον μου είναι να εξετάσω την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένω να καταθέσω και τροπολογίε, Αφόσον πιστεύω ότι επιδέχεται βελτιώσει η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις και τις αντιστάσεις και αντιδράσεις στο σχέδιο της Επιτροπής, αλλά για άλλους λόγους φαντάζομαι, όχι για τους λόγους ε, του κύριου Μαρτάν που είναι σελίδιν κατά της, ε, αναφαδόν μάλλον κατά της ε, εσωτερικής αγοράς. Οι υπόλοιποι φαντάζομαι θέλετε απλώς να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όχι να την καταργήσουμε παντελώς. Οπότε, μια και στόχος μας είναι η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να δούμε αν το προτινόμενο εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει και να είναι εύχριστο. Η κυρία Χάρκιν με ρώτησε γιατί ασχολούμαι με το θέμα της σιωπηρής ε, συνένεσης ή της σιωπηρής συγκατάθεσης. Αυτό το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση που οι αρχές της χώρας υποδοχής δεν έχουν αρνητική γνώμη, ε, τεκμέρεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις και άρα ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να αναπτύξει τις δραστηριότητες του. Αυτό θεωρείται ως σιωπηρή έγκριση ή σιωπηρή αποδοχή της λειτουργικότητας, εγκυρότητας της ηλεκτρονικής κάρτας. Οπότε αυτή η σιωπηρή έγκριση δεν ισχύει λόγω καθυστέρησης, ε, λόγω παρα... παρανόησης, για παράδειγμα ή λόγω έλλειψης αφήνειας. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν έχει νόημα η σιωπηρή αποδοχή ή συγκατάθεση. Προτιμώ, για να είμαστε σίγουροι για την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής κάρτας, να απαιτούμε ρητή έγκριση, ρητή αποδοχή, ρητή συγκατάθεση. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση στη διαδικασία έγκρισης η συγκατάθεση ή η έγκριση να είναι ρητή και όχι σιωπηρή ή απλώς να τεκμέρεται. Αλλιώς πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες για βελτίωση του κειμένου και περιμένω και τις προτάσεις των σκιωδών εισηγητών και των λοιπόν συναδέλφων. Σας ευχαριστώ, ήταν πραγματικά πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και νομίζω ότι και από χρονική άποψη είμαστε εντάξει γιατί η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λήγει στις 24 Οκτωβρίου άρα έχετε αρκετό χρόνο για δράσεις και για εκπόνηση τροπολογιών. Η εξέταση των τροπολογιών θα λάβει χώρα στις 20 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις αρχές Ιανουαρίου ή και κάπως αργότερα, ίσως τον Ιανουάριο. Οπότε έχουμε χρόνο, θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά πολύ διαφωτιστική ή και όχι. Σε κάποια σημεία ίσως η συζήτηση. Πάντως χρήσιμη ήταν. Η επόμενη μας συνεδρία θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου. πρωί και απόγευμα στις Βρυξέλλες. Αυτά. Καλό σας απόγευμα και καλά να περάσετε μέχρι τότε. Γεια σας.